Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στα ρωσικά. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Φροντίστε παρακαλώ να πάρει τα ακουστικά της η κυρία Αλεξιάγεβα, παρόλο που καταλαβαίνει αγγλικά. Συνεδριάζουν από κοινού η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που εκπροσωπείται εδώ από τον ε, πρόεδρο τη, κ. Αλμπερτίνη, η Επιτροπή Ανάπτυξη, που την εκπροσωπεί η Αντιπρόεδρο Στρίφλερ, και η Τρίτη Επιτροπή είναι η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκπροσωπείται εδώ από την υποφαινομένη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη αυτών των τριών επιτροπών στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Και επίσης έχουμε και την αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας που εκπροσωπείται από τον κύριο Φλέγκενστάιν τον πρόεδρό της. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε κυρίως πολύ πρακτικοί και να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τους βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ, να τους ξανασεχαρούμε. Ο κύριος Κοβάλιοφ μετά από ένα φρενήρες πρόγραμμα που είχε το τελευταίο διήμερο έμεινε να ξεκουραστεί λίγο άνθρωπος και μάλιστα είχα τη χαρά να συνοδεύσω από τη Μόσχα στο Στρασβούργο και με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα και στη Μόσχα σε μια διεθνή διάσκεψη για τη μνήμη του Αντρέη Ζαχάροφ. Μάλιστα η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ήταν η 40η επέτειος της, ε, του θανάτου του Αντζέι Ζαχάροφ που ήταν από τους ιδρυτές της οργάνωσης Memorial. Επί τη ευκαιρία εξέτασα και την κατάσταση στη Ρωσία, μια και βρέθηκα επί τόπου, και πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γεκάτερινμπορκ, στο κατόφλι της Σιβηρίας ουσιαστικά και μάλιστα εκεί συνάντησε έναν νεαρό ακτιβιστή, τον Αλεξέη Νικηφόροφ, 25 ετών, που κατά τη γνώμη μου ε, φυλακίστηκε παράνομα εξαιτίας ε, των πολιτικών του πεπιθήσεων και δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να ζητήσω από τους βραβευθέντες ε, με το βραβείο Ζαχάροφ να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ανησυχεί η επιδείνωση της κατάστασης για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε συγκλονιστεί από τις ειδήσει που ακούσαμε λίγο πριν αναλάβουμε τη θητεία μας, τη δολοφονία δηλαδή της Νατάλια Στεμίροβα. Βέβαια ακούσαμε με ικανοποίηση ότι η οργάνωση Memorial θα ε, ξαναναλάβει το έργο της και στο Βόρειο Κάφκασο, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλμπερτίνη, που είναι ο πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Αλμπερτίνη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Χάουταλα. Και εγώ θα ήθελα να πω ε, και να, μια, να απευθύνω θερμό, θερμή υποδοχή και να καλωσορίσω τους βραβευθέντες με αυτό το τόσο πολύτιμο βραβείο και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων. Ε, ελπίζω πως ε, θα σας βοηθήσει να ε, αναπτύξετε ακόμη περισσότερο την αφοσίωσή σας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στο In Memorial, αυτή τη, μη, τη ρωσική μη κυβερνητική, είναι μόνο μία πτυχή των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις επαφές με την Ρωσική Ομοσπονδία. Θα ήθελα να σας θυμίσω τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την, τις δολοφονίες ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ε, κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, την κατάσταση στον, στον Κάφκασο, τον Βόρειο, κυρίως στην Τσετσενία. Και θα ήθελα επίσης να θυμίσω τις ακροάσεις που έγιναν ε, στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές τελευταία το Σεπτέμβριο του 2009 όπου προείδρευσε η συνάδελφος Σάουταλα στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και όλα αυτά μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ρωσία, να διατυπώνουμε συστάσεις τόσο στο Συμβούλιο όσο και στην Κομισιόν για την ανάπτυξη των ε, καταλλήλων σχέσεων ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Εμείς Επίσης εκφράζουμε τι θέσει μας πριν από τις διασκέψεις κορυφής μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και παρακολουθούμε με προσοχή τις διαπραγματεύσει για τη νέα συμφωνία συνεργασίας που θα πρέπει να προβλέπει μεταξύ άλλων και μια σημαντική ανάπτυξη του συστήματος σεβασμού των ε, πολιτιακών δικαιωμάτων στην πρώην Σοβιετική Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί πως η στρατηγική εταιρική σχέση που θέλει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία θα πρέπει να βασίζεται σε ανθρώπινες αξίες. Γι' αυτό και το βραβείο έχει και αυτήν την βαθύτερη σημασία. Την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ένα βασικό κριτήριο των διμερών μας, των διμερών μας σχέσεων. Δηλαδή, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της νέας Συμφωνίας Συνεργασίας Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, θα θέλαμε ε, ειλικρινά να εκφράσουμε μεγάλο θαυμασμό για το θάρρος και την αποφασιστικότητα των εκπροσώπων του, της οργάνωσης Memorial και τον κύριο Ορλόφ, την κυρία Αλεξέγεβα, τον κύριο Κόβαλεφ που είναι παρόν μαζί μας ακόμα και αν ε, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Ε, εγώ θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς πιστεύετε πως το Κοινοβούλιο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει στον καθημερινό σας αγώνα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις δικέ σα μαρτυρίες, τις προτάσεις σας, για να τι υιοθετήσουμε και να τις διαβιβάσουμε, έτσι ώστε αυτή η εξαιρετική σας δουλειά, πολιτική και πολιτική δέσμευση που τόσο σας έχει κάνει να υποφέρετε, να μπορέσει να βρει μια σημαντική διέξοδο και να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αλμπερτίνη. Να ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Τρίφλερ, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Oui. Ως πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμά τους ε, υψηλούς προσκεκλημένους μας και χαίρομαι για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στην οργάνωση Memorial που εκπροσωπείται εδώ από τους καλεσμένους μας γιατί Συμβολίζει την αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θαραλέο αγώνα που δίνεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ω Επιτροπή ε, ανάπτυξη θα ήθελα να εκφράσω τον αμέριστο θαυμασμό μου για την οργάνωση Memorial και για το έργο της ε, στις ε, ζώνες σύγκρουσης και στις ένοπλες διαμάχες στη Ρωσία. είναι σημαντική πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να μπορέσει να δρομολογηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν χάσει οποιοδήποτε βιοποριστικό μέσο ή έχουν εκτοπιστεί εξαιτία μιας διένεξης. Μάλιστα, ο σεβασμό των στοιχειωδών ε, ανθρωπιστικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό παράγοντα για την προσπάθεια παρασυφιλία από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ένοπλη φάση τη διένεξη. Στις τελευταίες δεκαετίες είδαμε μια έξαρση της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ε, ε, εποχές και περίοδους σύγκρουσης. Έχουμε σοβαρή καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάλυση και ο αγώνας της οργάνωσης Memorial ε, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ανατροπή αυτής της τάσης. Λεπτομεριακές πληροφορίες και η διάδοσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αφυπνιστεί το κοινό και να δημιουργηθεί απαραίτητη πολιτική πίεση. Ε, ο εντοπισμό και η καταγγελία των ε, ενόχων ε, καταπολεμά το, την ατιμορρησία και αποτελεί μια επένδυση και για το μέλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Κοβάλ, κυρία Κοβάλεφ, κύριε, Κο, κύριε Ορλοφ, κύριε Αλεξία Γεφά, το έργο σας είναι ουσιώδες αλλά ταυτόχρονα έχουμε επίγνωση και το επικίνδυνο χαρακτήρα του. Σα διαβεβαιώνουμε για την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι θα σα δώσει κουράγιο και σε εσά και σε όλου του προσπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να συνεχίσετε την πορεία σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλά να, να σας πω ότι έχουν διανεμηθεί δύο κείμενα. Είναι τα ανακοινωθέντα τύπου, το χθεσινό, Human Rights Resumes Work in Chechnya και ένα άλλο έγγραφο πολύ σημαντικό είναι ένας κατάλογος συστάσεων από ΜΚΟ που οι περισσότερες είναι ρωσικές πριν από τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Στοκχόλμη τον Νοέμβριο. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε και αυτό να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ορλόφ για πέντε λεπτά περίπου. Και μετά στην κυρία Λεξέγεβα. Κύριε Ορλόφ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι που μου δίνετε το λόγο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την βράβευσή μας με το βραβείο Ζαχάροφ καθώ και για τα εγκάρδια λόγια που μας απευθύνατε πριν από λίγο. Άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Βέβαια, αυτό θέτει και ένα ερώτημα Γνωρίζετε σίγουρα ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία δεν είναι ικανοποιητική και ότι μάλλον επιδεινώνεται. Ακόμα περισσότερο πριν από λίγα χρόνια σημειώνονταν συχνά βαριές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι και σε εμά, δηλαδή στι οργανώσει ανθρώπινων δικαιωμάτων, σημειώνονται πιέσει. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει περιπτώσεις φόνων υπερασπιστών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην περιοχή του Καυκάσου και αλλού. Γι' αυτό το λόγο Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται βοήθεια η κίνηση προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται η Ρωσία να παρεκκλίνει από το δρόμο της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Εάν συγγύσουμε εμείς, οι ελπίδες θα μειώνονται όλο και λιγότερο να επιστρέψει η Ρωσία στον σωστό δρόμο. Σε ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γνωρίζετε ποια μορφή έχει λάβει ο διάλογος αυτός. Διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δύο φορές τον χρόνο. Ως οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμείς παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό τον διάλογο αυτό σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνάντηση που διεξάγεται, παρακολουθούμε, συντάσσουμε εκθέσεις. Μετά όμως τι γίνεται. Η διαβούλευση αυτή, οι διαβουλεύσεις αυτές για μας είναι στην ουσία κούφιες, χωρίς περιεχόμενο. Προσέρχονται δηλαδή σε αυτές αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιωματούχοι από τη Ρωσική πλευρά και συζητούν η ευρωπαϊκή πλευρά θέτει ορισμένα ερωτήματα και η ρωσική πλευρά απαντά ορισμένες φορές με ψεύδι, ορισμένες φορές με διάφορες ιστορίες και βλέπουμε ότι εν τέλει ικανοποιείται με τις απαντήσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ήταν εν τέλει όλο το αποτέλεσμα του διαλόγου. Δέχονται δηλαδή οι Ευρωπαίοι κάποιες, κάποια ψεύδιος απαντήσεις και εν τέλει συμφωνούν να ξανασυναντηθούν μετά από έξι μήνες. Δεν είναι πραγματικός διάλογος αυτός. Αλλάζει πάλι η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται άλλοι οι οποίοι οργανώνουν και συνεχίζουν τον διάλογο. Και τα ερωτήματα που είχαν τεθεί στην πρώτη φορά στον πρώτο διάλογο δεν επανέρχονται στον επόμενο προχωρούν σε διαφορετικά θέματα. Σε αυτούς τους διαλόγους δεν συμμετέχουν οι μη κρατικέ οργανώσεις, διότι η Ρωσία απορρίπτει τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι μέγα μείον για τον, για την αξία του διαλόγου, διότι εν τέλει μόνο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι αυτοί οι οποίοι συνέρχονται εκεί και συζητούν. Και συχνά λένε, α, δεν ξέρουμε ήδη ότι δεν είμαστε ειδικοί. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιμείνει να περιληφθούν στις διαβουλεύσεις αυτές εμπειρογνώμονες από τις οργανώσεις, από τις μη οργανώσεις, από τα δικαστήρια, και να μην δέχεται το όχι των ρωσικών αρχών. Οι δεμοί, οι διάλογοι αυτοί στερούνται νοήματος. Εάν δηλαδή στους διαλόγους δεν συμπεριλαμβάνονται και άλλες πλευρές της κοινωνίας. Μπορούμε εμείς να συντάσσουμε εκθέσεις, αλλά δεν ωφελεί σε τίποτα. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν υπεύθυνοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χειρίζονται τα, τα των διαλόγων αυτών. Αλλά προχωρούν χωρίς να σκέφτονται αρκετά τα πράγματα. Χρειάζεται να εξευρεθούν νέοι τρόποι, νέες μορφές των διαλόγων αυτών. Και η ρωσική πλευρά πρέπει να διαβουλευτεί μετά του οίκου της, αλλά μέχρι τώρα το απορρίπτει αυτό. Και αυτό βέβαια επηρεάζει ολόκληρη την διαβούλευση. Καλά θα ήταν να προσέρχεται στην ε, Ρωσία μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη πριν από την εξαγωγή του διαλόγου για να αναζητήσει εκεί τις αληθινές απαντήσεις στα ερωτήματά της. Το σημαντικό επίσης, όπως είπα, είναι να μπορούν να συμμετέχουν και οι μη κρατικέ οργανώσεις. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, στα οποία απαντά η Ρωσία αμέσω αρνητικά. νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβάλει επαρκείς προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι ο διάλογος αυτός θα έχει κάποια αξία. Αν είναι έτσι, μπορούν να καταργηθούν οι διαβουλεύσεις αυτές, διότι δεν έχουν νόημα. Καλύτερα να μην γίνονται καθόλου, εάν να γίνονται έτσι οι διαβουλεύσεις αυτές. Και νομίζω ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν στη νέα συμφωνία συνεργασίας και να έχουν και σημαντική θέση εντός αυτής. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος των μη κρατικών οργανώσεων να απευθύνεται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητεί να ενταχθεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Συμφωνία Συνεργασίας αφού είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Όμως δεν έγινε τίποτα διότι η Ρωσία αντιστέκεται. Το ερώτημα που θέτω λοιπόν είναι τι νόημα έχει τότε αυτή η συμφωνία, η νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν από αυτήν θα αφαιρεθεί ένα σημαντικό μέρος. ενώ θα έπρεπε να είναι ένα σημαντικό μέρος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκαλούνται αμφιβολίες σε εμά, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλαίσια του διαλόγου με τη Ρωσία είναι πραγματικά διατεθειμένη να δώσει την απαραίτητη προσοχή στα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ένα τελευταίο. Σας ευχαριστούμε που επιτρέψατε να καταθέσουμε εδώ τις συστάσεις μας, ξεκινώντας από την διάσκεψη της Στοκχόλμης. Έρχομαι στην απειλή κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βόρειο Καύκασο έχουμε με τις συστάσεις μας τονίσει ότι χρειάζεται να δοθεί βοήθεια στην κοινωνία των πολιτών εκεί. Εδώ πρέπει να υποστηριχθεί η Ρωσία, διότι νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη τη Ρωσία. Η κυρία Χαουτάλα, σας ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Γνωρίζω ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν νέε μορφέ για τι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί όλοι είμαστε απογοητευμένοι για το γεγονό ότι δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί μπορούμε να συνεργαστούμε και με εσά πράγματι. Τώρα αυτή η διαδοχική προεδρία. Έχουμε τώρα την ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής. Άρα θα υπάρξει ένα νέο είδος συνέχειας. Και εμείς εδώ, οι Ευρωβουλευτές, ελπίζουμε πολύ ότι θα αποδώσει αυτή η συνέχεια στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι εδώ ανοίγεται μια ε, σημαντική ευκαιρία θα μπορέσουμε ίσως να θεσπίσουμε νέες πρακτικές. Παρακαλώ η κυρία Αλεξέγεβα, 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Εστερνίζομαι πλήρως αυτά που είπε ο κύριος Ορλόφ. Με διευκόλυνε πολύ. Δεν χρειάζεται καν να εξαντλήσω το επτάλεπτο. Και χαίρομαι που ήδη υπάρχουν και κάποιες συστάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πολύ συγκεκριμένες πτυχές προκειμένου να βοηθήσουμε τους ακτιβιστές μας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να συνδράμουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτον, σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε την αίσθηση ότι οι ακτιβιστές μας ε, τελούν υπό απειλή. Στο Βόρειο Κάφκασο, για παράδειγμα, στην Τσετσενία, στην Ιγκουσετία, τον Ταγκεστάν. Εκεί απειλείται η ζωή των ανθρώπων αυτών. Παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να διευκολύνουμε τη χορήγηση θεωρήσεων. Να τους δίνουμε πολύ πιο εύκολα βίζες ώστε να μπορούν ανα πάσα στιγμή να εγκαταλείψουν τη χώρα. Μάλιστα πολλοί δεν ζητούν καν θεωρήσεις για τους εαυτούς τους αλλά για τις οικογένειές τους. Και πολύ συχνά δεν δολοφονεί το ίδιο ο δημοσιογράφο ή ο ακτιβιστή, αλλά ένα μέλο τη οικογένειά του, ένα συγγενή του, κάποιο που αγαπάει πολύ. Δεν υπάρχουν ασφαλεί, ασφαλείς τοποθεσίες για τους ανθρώπου αυτούς στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν μπορούν να πάνε στη Μόσχα και να κρυφτούν. Οπουδήποτε η ζωή τους κινδυνεύει. Γι' αυτό σας θερμοπαρακαλώ διευκολύνεται τη χορήγηση θεωρήσεων για τους ανθρώπους αυτούς. Λάβετε μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και οι συγγενείς τους και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δρούν στην περιοχή και τα μέλη τους να μπορούν εύκολα να φύγουν από τη χώρα και να λαμβάνουν πολύ πιο εύκολα βίζες και οι ίδιοι και οι συγγενείς τους, τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ένα δεύτερο αίτημα θα ήθελα να απευθύνω προς την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εξαιτίας ε, και της σοβούσας κρίσης Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου που ελοχεύει στην περιοχή. Κάτι τέτοιο γίνεται ήδη στην Ιγκουσιατία και το Ταγκεστάν. Θα σας θερμοπαρακαλούσα λοιπόν ιδιαίτερα την Επιτροπή Ανάπτυξης να εκπονήσετε κάποια προγράμματα για να διευκολυθούν οι νέοι της περιοχής του Καυκάσου, να δημιουργηθούν ευκαιρίες ε, για κατάρτιση ή απασχόληση. Δεν λέω ότι όλοι είναι τρομοκράτες, όλοι οι άνεργοι είναι τρομοκράτες, αλλά αν το 80% του πληθυσμού είναι άνεργοι, τότε δημιουργείται μια με κατάσταση και πρόσφορο έδαφος ε, για μισαροδοξία, θρησκευτικό φανατισμό και τρομοκρατία. Και εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση, εγκρίνοντας κάποια προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ή δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους αυτούς για να σπουδάσουν ή να εργαστούν και να βελτιωθεί το βιωτικό τους επίπεδο. Έτσι θα μειωθεί και η απειλή της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά τη Χάιντι Χάουταλα που επισκέφθηκε στη φυλακή τον Αλεξέη Νίκοροφ. Ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή. Και αν γνωρίζετε και άλλες περιπτώσεις ε, φυλακισμένων, θα μπορούσατε να οργανώσετε πολλές τέτοιες επισκέψεις στις φυλακές, όπου ευρωβουλευτές θα επισκέπτονται ε, φυλακισμένους ε, για λόγους συνείδησης. Όχι μόνο ευρωβουλευτές, αλλά και, άλλοι, και άλλες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι που περιμένουν τη δίκη τους. Δυστυχώς ε, τα δικαστήρια που υποτίθεται είναι ανεξάρτητα λαμβάνουν ε, πολιτικές αποφάσεις και χειραγωγούνται οι δικαστές από τους πολιτικούς. Οπότε αν ε, επισκεφθείτε τέτοιους πολιτικούς κρατούμενους, ακόμη και στη φάση της προσωρινής τους κράτησης πριν τη δίκη θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ο Αντρέι Σόκολοφ ε, που κρατείται στο Γεκατέρινμπουργκ είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθη ε, με ψευδείς κατηγορίες. Έγινε μια σκευωρή βάρος του και συνελήφθη παρόλο που το έργο του ήταν πολύ αποτελεσματικό. Μάλλον επειδή το έργο του ήταν πολύ αποτελεσματικό, Σας ε, παροτρύνω λοιπόν να επισκεφτείτε τον, Άντρε, τον Αλέξη Σόκολοφ πριν δικαστεί, γιατί με μια τέτοια επίσκεψη ίσως ασκηθεί πίεση και αλλάξει η απόφαση, μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο του. Γνωρίζετε τους ε, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι και τον Μιχαήλ Έπιτιφ. Πραγματικά εκεί στις ε, δικές τους δίκες γίνεται κάτι τελείως παρανοϊκό και αλλοπρόσαλο είναι τόσο εμφανής η παραποίηση ε, των στοιχείων, των αποδεικτικών στοιχείων, που οποιαδήποτε επίσκεψη προσωπικότητας ε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα τους βοηθήσει πολύ. Οποιαδήποτε διεθνής παρουσία στη δίκη τους θα βοηθήσει πολύ και ίσως ε, μειωθεί η πιθανότητα μιας άδικης ανελαίτης και μακροχρόνιας ποινής. Σας ζητώ συγγνώμη που έχω ένα τόσο μακροσκελή κατάλογο ετοιμάτων, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας όσο γίνεται. Ευχαριστούμε κυρία Αλεξέγεβα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και τέτοιες νομοθετικές διατάξεις ε, που ισχύουν στη Ρωσική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα τις παραγράφους ε, στον ε, ποινικό κώδικα για τις ε, δραστηριότητες των εξτρεμιστών. Το άρθρο 282, δεν κάνω λάθος, του ποινικού κώδικα. Πολύ φυλακισμένοι που συνάντησα ανησυχούν για τη νέα μονάδα στο Υπουργείο Σωτερικών, το Center E, που πραγματικά ασκεί αφόρητες πιέσεις στους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω ένα εκτενή κατάλογο ομιλητών. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω τον κύριο Φλέκεσταϊν αν θέλει να λάβει το λόγο και μετά μια κυρία ο πρόεδρος αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Ρωσία και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Κέλλαμ την κυρία Λόμπιχλερ και άλλους. Μετά τον κύριο Φλέκεστάιν, καλό θα είναι οι ομιλητές να μην ξεπεράσουν το δίλεπτο. Έχετε το λόγο κύριε Φλέκεστάιν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με τη σειρά μου επιθυμώ να συγχαρώ τους εκπροσώπους του μεμορίαλ για την βράβευσή τους και προσθέτω ένα λόγο ακόμη. Για πολλά χρόνια ήσασταν το σύμβολο μιας μη κρατικής οργάνωσης και με τον τρόπο αυτό δώσατε θάρρος και σε πολλούς άλλους να αναλάβουν παρόμοιο έργο με το δικό σας. και γι' αυτό το λόγο σας αξίζουν οι ευχαριστίες μας. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται οι κοινωνίες της Ευρώπης και τις οποίες επικαλούνται συχνά. Για τον λόγο αυτό οι αξίες αυτές οφείλουν να διέπουν την καθημερινή μας εργασία στην Ευρωβουλή. Τίθεται το ερώτημα πώς εμείς ως Ευρωβουλευτές μπορούμε να πείσουμε τους Ρώσους εταίρους μας ότι χρειάζεται να κάνουν την αντιπαράθεση, την αντιμετώπιση του στελνικού παρελθόντος και ότι το χτίσιμο μιας αλληλέγγυας κοινωνίας με ανθρώπινα δικαιώματα δεν οδηγεί στην αποδυνάμωση του κράτους. Αντίθετα, ενισχύονται οι κρατικές δομές με τον τρόπο αυτό. Εμείς θέλουμε μια θετική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Αλλά θέλουμε στην Ήπειρο αυτή να υπάρχει ένα σταθερό και ειρηνικό μέλλον. Σε αυτή την εταιρική σχέση πρέπει, αυτή μάλλον εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται σε διαφάνεια και ειλικρίνεια. Μόνο μαζί με κοινή συνεργασία μπορούμε να χτίσουμε ένα τέτοιο μέλλον. Χρειάζεται όμως μια εταιρική σχέση που να βασίζεται σε εμπιστοσύνη και σε κοινέ αξίες που να διέπουν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους Ρώσους εταίρους να διδαχθούν από τις δικές μας εμπειρίες που δεν ήταν πάντοτε θετικές. Οφείλουμε να δεχθούμε ότι κάθε χώρα θα βρει το δικό της τρόπο να ιδρύσει μια κοινωνία που να λειτουργεί. Και χρειάζεται υποστήριξη οργανώσεων όπως η Memorial. Κύριε Ορλόφ, μετά από τη δική σας παρέμβαση οφείλω να πω ότι έχετε δίκιο στις συζητήσεις που θα κάνουμε και που θα κάνει και η αντιπροσωπεία για σχέση με τη Ρωσία πρέπει να επανερχόμαστε διαρκώς στο θέμα και όχι να θεωρούμε ότι έχει λήξει. Τον Ιανουάριο όταν θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους μας της Ρωσικής Δούμα θα αναφερθούμε ρητά στο θέμα του βραβείου Ζαχάροφ του 2009 και έχουμε περιλάβει και ειδικό θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Ο Βέρνερ Σούλτς, συναδελφός μας, θα κάνει τη σωστή προπαρασκευή και θα διεξαγάγει τη συζήτηση με τρόπο που να μην ολοκληρωθεί, μην λήξει η συζήτηση αυτή όταν θα λήξουν οι εργασίε μα, αλλά αντίθετα θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα συνεργασία με του Ρώσου βουλευτέ, ώστε του χρόνου, τον Μάιο κατά πάσα πιθανότητα, να διεξαγάγουμε μια συνεδρίαση μονάχα για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και θα δούμε, θα φροντίσουμε ώστε στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης να μπορέσουν να διεξαχθούν συζητήσεις και με εσά και με άλλους που εργάζονται δραστήρια υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην γίνουν συζητήσεις με το Memorial, με την Διεθνή Αμνηστία κτλ. Έχετε δίκιο λοιπόν όταν λέτε ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να επιμείνουμε περισσότερο, να μην διατηρήσουμε σχέσεις και επαφές μοναχά με τις επίσημες αρχές, αλλά και με ανθρώπους όπως εσάς. Και σας βεβαιώ ότι για τα επόμενα 5 ή 4,5 τέλος πάντων χρόνια θα το πράξουμε. Ένα τελευταίο θέμα. Νομίζω ότι στις συζητήσεις μας με τους Ρώσους εταίρους μας θα μπορούμε να αναμένουμε κάποιε πρόοδου μόνο εφόσον του δείξουμε την τον απαραίτητο σεβασμό. Δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συζητήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε οι μεν τους δε ώστε να βαδίσουμε σε ένα καλύτερο δρόμο. Και αυτό προφανές, προφανώς είναι δύσκολο καμιά φορά να επιτευχθεί, να βρεθεί δηλαδή ο σωστός δρόμος. γιατί μόνο τότε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και εσάς και άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Σας ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν. Το λόγο θα λάβει η κυρία Λόχ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τους βραβευθέντες για το έργο που έχουν επιτελέσει στη Ρωσία. Θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Σογκλόφ για τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα τον ευχαριστήσω για τις συγκεκριμένε προτάσεις του. Παρόμοια κριτική ακούσαμε και στην ακρόαση που διεξαγάγαμε για την Κίνα ότι ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδίδει πολύ περιορισμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Ας μην απατώμεθα. Οι διάλογοι αυτοί έχουν ως στόχο να περιορίζουν τη δημόσια κριτική. Θα ήταν βέβαια παράλογο να είναι κανείς κατά του διαλόγου, αλλά και η διεξαγωγή διαλόγου χωρίς αποτελέσματα είναι στην ουσία απάτη και αυταπάτη. Και δεν την πιστεύει πια η κοινωνία των πολιτών σε καμία από τις συμμετέχουσες χώρες. Έχω μια ερώτηση. Ο πρόεδρος Μετβιέντεφ ζήτησε αναθεώρηση πρότεινε αναθεώρηση του καθεστώτος των ε, μη κρατικών οργανώσεων στη Ρωσία. Νομίζετε ότι θα γίνει αυτό γιατί δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Τώρα η κυρία Αλεξέγευνα που εξήγησε ποια βοήθεια χρειάζονται οι περασπιστές ε, υπερασπίστες των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι χώρε μέλη με υποστήριξη τη Ένωση, να συντάξουν προγράμματα που να επιτρέπουν να εξέρχονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οικογένειές τους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο γρήγορα και μη γραφειοκρατικά. Αντί να μην περνούν δηλαδή μήνες και χρόνια μέσα σε περίπλοκες διαδικασίες ασύλου. Είναι πραγματικά κατανόητο πως χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαναστέλνουν πίσω στη Ρωσία ανθρώπους που έχουν έρθει για παράδειγμα από την Τσετσενία επειδή αρνούνται να αντιληφθούν πόσο δύσκολα και επικίνδυνα, δύσκολη και επικίνδυνη είναι η κατάσταση εκεί. Και εσείς κύριε Αλεξέγεβα εξηγήσατε τελευταία ποια είναι τα ισχυρά και λιγότερο ισχυρά σημεία της ρωσικής κοινωνίας. Εσείς μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα πράγματα, εκτός βέβαια από τις απειλές, δεν είναι μόνο οι απειλές δηλαδή, που ε, καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόχ Μπίλερ. Θα διαβάσω τον κατάλογο των αγορητών για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Θα ακούσουμε μερικές ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Αλεξέγεβα και τον κύριο Λόφ και μετά θα έχουμε το δεύτερο γύρο. Μήπως παρέλειψε κανένα από τον κατάλογο? Α, τον κύριο Πέτερλε. Δεν πειράζει, γιατί Κάποιος με πρόλαβε και διατύπωσε την ερώτησή μου. Μπράβο, σας ευχαριστούμε για την γενοδορία σας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Τουνακέλα, μετά στην κυρία Στρίφλερ και θα ακούσουμε μετά τους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Κέλαμ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έζησα πάνω από 40 χρόνια στην Ευρωσοβιετική Ένωση και καταφέραμε να ξεφύγουμε από την ε, Σοβιετική Ένωση και να ανακτήσουμε την ελευθερία μας, αλλά έχουμε κοινέ ελπίδες, κοινό πεπρωμένο και θέλουμε να στηρίξουμε τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ και η επίσκεψη των βραβευθέντων εδώ, ιδιαίτερα για μένα. Θα ήθελα να αναφέρω μία παράγραφο από τη χθεσινή ομιλία του Σεργέη Κοβάλιοφ, μίλησε για την συνεισφορά της Ρωσίας στα ανθρώπινα δικαιώματα από τα τέλη της δεκαετίας του 60 για τη διαμόρφωση της νέας πολιτικής παιδείας στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται ουσιαστικά μόνο για τη Ρωσία, αλλά για την κοινή μας κληρονομιά και τις κοινέ μας ευθύνες. Και υπήρχαν κάποιοι σοβιετικοί προσπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινητοποίησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη που την αφύπνισαν. Και όπως είπε και ο Σεργέη Κοβάλιοφ, οι δυτικοί ηγέτες, χάρη στην κινητοποίηση αυτή, άλλαξαν γνώμη. Γιατί οι δυτικοί ηγέτες δεν ήταν προετοιμασμένοι για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή ήταν λοιπόν η συμβολή της των Σοβιετικών και Ρωσικών Οργανώσεων Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το πιο ανησυχητικό πάντως σήμερα πράγμα είναι η κατάσταση στο Βόρειο Κάφκασο. Γιατί κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απελπιστεί. δεν τρέφει πια καμία ελπίδα για βελτίωση της κατάστασης στο Βόρειο Κάφκασο. Και όπως αναφέρθηκε, οι φίλοι μας εκεί έχουν ε, μείνει μόνοι τους, εγκαταλελειμμένοι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που υψώνουν τη φωνή τους και προσπαθούν ε, να ζητήσουν τη δίωξη των ενόχων. Και μάλιστα μερικοί που διεκδίκησαν τέτοια δίωξη των ενόχων έχουν ήδη δολοφονηθεί. Τιμωρούνται οι αθώοι, ενώ οι ένοχοι μένουν ατιμόρυτοι. Αυτό το θέμα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας απασχολήσει. Δεύτερο, πόσο σοβαροί είμαστε με τι σοβαρότητα πραγματικά αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί είναι κοινό καθήκον και ευθύνη μας να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ε, εύρωσης και υγιούς κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Δεν μπορούμε να ευημερίσουμε στην Ευρώπη αν δεν εξασφαλίσουμε μια πραγματικά και γνήσια δημοκρατική Ρωσία η Ρωσία φαίνεται να μεταχειρίζεται ακόμη τους παλιούς σοβιετικούς τρόπους αντιμετώπισης των πραγμάτων. Οι Ρώσοι ηγέτες προσποιούνται ότι έχουν δημοκρατία επειδή υπάρχουν κάποιοι θεσμοί. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσποιούνται ότι πιστεύουν τη Ρωσία. Το αναφέραμε αυτό, το έχουμε επισημάνει. Και το όλο θέμα, όπως είπαν οι φίλοι μας, αφορά την ευρωπαϊκή σοβαρότητα και την ε, πραγματική δέσμευση υπέρ της αλλαγής. Πολλά αναφέρθηκαν για, τα, για τους θελάμους αερίου στο ναζιστικό καθεστώς. Σήμερα υπάρχουν άλλοι τρόποι, αλλά δυστυχώς ε, ακόμη και σήμερα καταπατάται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και φημώνεται η ασφικτιά στη, στη ροή αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Η πρότασή μου είναι εξή. Όπως αναφέρθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαινίασε τη θητεία του την εποχή που δολοφονήθηκε η Νατάλια Στεμίροβα. Λοιπόν, δίκιο θα ήταν να θυμηθούμε τη μνήμη της και να της αποτίσουμε φόρο τιμής δίνοντας το όνομά της σε μια αίθουσα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πολύ σοφά μιλήσατε κύριε Κέλαμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Στρίφλερ και μετά στους καλεσμένους μας. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Ορλόφ, γιατί ορισμένα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και θα μπορούσαν να καταδείξουν δυσλειτουργίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβουλεύσει μαζί σας και με την οργάνωση Memorial πριν ξεκινήσει το διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Και αν ναι, υπάρχει συνέχεια μετά το διάλογο αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει συνέχεια και ανταλλαγή απόψεων, γιατί να κάνουμε τέτοια σχέδια και προγραμματισμό αν δεν υπάρχει πραγματικά ανταλλαγή απόψεων. Είναι ματαιοπονία. Και θα ήθελα να πω κάτι προς την κυρία Αλεξέγεβα. Όντως ε, θα πρέπει να επισκεφτούμε φυλακισμένους και κρατουμένους συνείδησης. Όταν ε, οι αντιπροσωπείς μας πραγματοποιούν επισκέψεις, ε, δεν ξέρω, πηγαίνουμε στις φυλακές, συναντιόμαστε με φυλακισμένους ή απλώς έχουμε συνεδριάσεις. Αυτά τα δύο σημεία, κατά τη γνώμη μου, είναι κέρια σημασίας για να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί σε όλα τα προγράμματα και σχέδια που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Στρίφλερ. Το λόγο έχει και πάλι ο κύριος Ορλόφ. Πόσα λεπτά. Όπως θέλετε. Τρία, τέσσερα λεπτά. Первое. Э, вот в ответ на ваш вопрос. Э, να απαντήσω πρώτα στην ερώτησή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβολεύεται μαζί μας πριν από τους διαλόγους. Και μετά, συνήθως, ο πρέσβης της χώρας που την Προεδρία έρχεται και μας αναπτύσσει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Αυτά που συζητούμε εμείς ελπίζουμε βέβαια μετά να μπουν στο διάλογο. Και ελπίζουμε να δοθούν και σοβαρές απαντήσεις σε σοβαρές ερωτήσεις. Κάθε φορά όμως διαπιστώνουμε ότι οι ελπίδες μας διαψεύδονται. Κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Τώρα είναι κάτι άλλο σημαντικό που είπατε. δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα στη χορήγηση υποστήριξη και στην άσκηση πίεση στη Ρώσικη Ομοσπονδία. Βέβαια πρέπει να υπάρχει σεβασμός και υποστήριξη, αλλά χρειάζεται μια ισορροπία. Χρειάζεται και η πίεση, αλλιώς δεν γίνεται. Δυστυχώ, εάν δεν ασκηθεί πίεση, δυστυχώ λέω, οι εκπρόσωποι της χώρας μου θα προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση για θέματα δημοκρατίας. Θα πούν ωραία λόγια, αλλά στην πραγματικότητα θα κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Στη Ρωσία δεν λειτουργούν σωστά οι εκλογές, δεν συζητεί πραγματικά το κοινοβούλιο. πρέπει να αναζητήσετε και να βρείτε συνομιλητές οι οποίοι πραγματικά να εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Πέραν των κυβερνώντων κομμάτων. Και είναι σωστό να βρείτε και το σωστό τρόπο να μιλήσετε με τους Ρώσους βουλευτές και να προσπαθήσετε να πείσετε τα πρόσωπα αυτά ότι η δημοκρατία είναι προς το συμφέρον εν τέλει και της Ρωσικής Βουλής. Και ότι δεν επιτρέπεται να δέχονται όσα υπαγορεύει μόνο το Κρεμλίνο. Οι αποφάσεις του Κρεμλίνου είναι αντιδημοκρατικές. Είναι σημαντικό και το κυβερνών κόμμα κάποια στιγμή να ξυπνήσει αλλά για την ώρα, όπως είπα, δεν διαγράφονται πολλές ελπίδες. Και ένα τελευταίο. Η δημοσιότητα. Η απήχηση στην κοινή γνώμη. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη, διότι στη Ρωσία ουδής γνωρίζει περί των διαλόγων αυτών. Κανένας δεν γνωρίζει ποιε είναι οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα δεν γνωρίζει τι, συζητούνται, ποια πράγματα συζητούνται. Τίποτα δεν φτάνει μέχρι την κοινή γνώμη. Εκεί πρέπει να φροντίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκύψει συγκεκριμένα στα θέματα αυτά. Και αυτά να τα θέσει στο διάλογο με τη Ρωσία. Για τον Κάφκασο. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω και άλλα στοιχεία για όποιον ενδιαφέρεται. Οι πρόσφυγες από την Τσετσενία οι οποίοι ζουν σε συνθήκες που είναι απειλητικές για τη ζωή τους να μπορούν να εξέρχονται διότι οι πρόσφυγες από την Τσετσενία δεν είναι και πραγματική Τσετσένοι στη χώρα τους. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείπουν τη χώρα. Όποιος πραγματικά απειλείται, όποιο κινδυνεύει η ζωή του δεν επιτρέπεται να ξαναστέλνεται στη Ρωσία. Αυτά ήθελα να πω. Thank ευχαριστώ. Ακούσαμε σήμερα στα Πόλωνο-Λευκορωσικά σύνορα εκατοντάδες τσετσένοι πρόσφυγες βρίσκονταν σε κατάσταση τραγική και διαμαρτύρονταν. Τώρα απειλούνται με κυρώσεις. Και δυστυχώ η πολιτική που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ προβληματική γιατί εικάζουμε ότι όλες οι χώρες έχουν αξιοπρεπείς, εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες αλλά δυστυχώς δεν ισχύει και τις, ε, τους αποθούμε προς την πρώτη χώρα εισόδου όπως είναι η Πολωνία. Έχουμε εκατοντάδες πάντως ε, τεζένους πρόσφυγες που σωρεύονται στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Κυρία Αλεξέγεβα, θα προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ειλικρινά, θα ήθελα να πω ότι μπορεί να μην κατάλαβα απόλυτα τις ερωτήσεις, γι' αυτό και ίσως να μην σας ικανοποιήσουν οι απαντήσεις μου. Ρωτήσατε για τους πρόσφυγες, κατά πώς θα πρέπει να γίνονται δεκτοί και μετά να επαναπροωθούνται. Δεν ήταν αυτό αυτό που είπα εγώ. Εγώ είπα ότι έχουμε συναδέλφους μας στην ε, Τσετσενία, στην Ιγκουσετία, στον Τακιστάν που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Στην ε, Ιγκουσετία για παράδειγμα είχα πάει πριν από ένα χρόνο και συνάντησα το Σαρίμπαλ Σεφ που μου είπε αμέσως μετά τη δολοφονία του Μαγκομέταρλο Μου είπε λοιπόν ότι πίστευε ότι πρώτα θα έχανα εγώ την ζωή μου, μετά ο Μαγκαμέτ και μετά ο κύριος Γευλόφ. Αλλά τελικά πρώτος δολοφονήθηκε ο Γευλόγεφ. Δεν ξέρουμε όμως ποιος θα είναι ο επόμενος. Και τελικά ο Μαξάριφ ήταν το δεύτερο θύμα. Μόνο εγώ και ο Μαγκαμέτ ε, βρισκόμαστε ζωή και πιστεύω ότι η ζωή του Μαγκαμέτ απειλείται σοβαρότατα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό. Πήγε πρώτα στη Φιλανδία, μετά στη Γαλλία, κατόπιν στι Ηνωμένε Πολιτείε και λέει ότι θέλει να επιστρέψει στη Τσετσενία, ότι η ζωή του δεν έχει νόημα μακριά από την Τσετσενία. Προσπαθώ να τον πείσω να παραμείνει στο εξωτερικό, αλλά εκείνος επιμένει, επιμένει να επιστρέψει και δεν μπορώ να τον μεταπίσω. Και υπάρχουν πολλές γυναίκες στην Τσετσενία που ε, δίνουν μάχη χρόνια ολόκληρα και λένε ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, γιατί η ζωή τους δεν έχει νόημα μακριά από την Τσετσενία. Και προτιμούν να δολοφονηθούν παρά να φύγουν και να εγκαταλείψουν τους συζύγους τους, τις οικογένειές τους, τη ζωή τους. Όλοι οι συγγενείς τους φοβούνται για τη ζωή τους και μάλιστα πολύ σωστά και εύλογα γιατί δεν ξέρουν πότε θα χάσουν τη ζωή τους ή πότε θα δολοφονηθούν οι συγγενείς τους. Ε, γίνονται δολοφονίες μελών της οικογένειας για εκφοβισμό των ακτιβιστών. Μου είπαν λοιπόν, ίσως εσείς ε, θα μπορούσατε να ζητήσετε ε, βίζα για να φύγουν οι οικογένειές μας από την Τσετσενία. Εμείς όμως θα παραμείνουμε και θα συνεχίσουμε το έργο μας. Φυσικά, ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για την ζωή του. Έτσι βέβαια κινδυνεύουμε να χάσουμε του ακτιβιστέ μα, του μαχητέ μα στην Τσετσενία. Πάντω, όταν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, προσπαθώ να του πείσω να φύγουν και να του διευκολύνω για να φύγουν. Αν θέλουν όμω να επιστρέψουν, δεν μπορώ να του εμποδίσω. Είναι ενήλικε και υπεύθυνα άτομα και θα αποφασίσουν για τον εαυτό του. Εφόσον όμω θέλουν να προστατεύσουν τι οικογένειε του, σα θερμοπαρακαλώ, σα εκλυπαρώ, κάντε κάτι για τι οικογένειε του, γιατί το αξίζουν. Οι, οι ίδιοι κινδυνεύουν βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Σώσουμε τουλάχιστον τις οικογένειές τους. Yes. Well, thank you, Mrs. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αλεξέιεβα. Νομίζω πως πρέπει να σκεφτούμε τα όσα είπε η κυρία Λόχμπιλερ στην παρέμβασή της, ότι δηλαδή θα πρέπει να, ρυθμίσουμε, να οργανώσουμε προγράμματα υποδοχής, όχι οπωσδήποτε να πάρουν άσυλο, αλλά να έχουν μια βίζα και να μπορούν να δουλέψουν σε μια χώρα της Ένωση για κάποια περίοδο όταν χρειάζεται. Και η Τσεχική Προεδρία πριν από την σημερινή Προεδρική, ε, ειδική με συγχωρείτε, ε, ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Η δική μας υποεπιτροπή εργάζεται για κάποιες τέτοιες ιδέες για το πώς θα αναπτύξουμε καλύτερους μηχανισμούς ώστε να στηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια ιδέα την οποία ναι, θα εξετάζουμε. Τώρα, οι εξή ε, ομιλητέ είναι στο διάλογο μου. Ο χρόνο είναι περιορισμένο. Όλοι θέλουν να δείξουν αλληλεγγύη. Μπορείτε να μιλήσετε για λιγότερο από δύο λεπτά. Και αν έχουμε χρόνο, ο, ο άλλος ένας ομιλητής και οι καλεσμένοι μας, ο κύριος Στάλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αλεξέγεβα, κύριε Ορλόφ. Θα ήθελα προσωπικά να σας καλωσορίσω. Το βραβείο Ζαχάραφ που σας απονομήθηκε και η σημερινή σας παρουσία εδώ αξίζουν πολύ περισσότερα από 10, 15, 20 επισήμους διαλόγους με τις επίσημες ε, ρωσικές αρχές. Γιατί αξίζουν περισσότερο, γιατί εδώ βλέπουμε πραγματικά ποια είναι η σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα δικαιώματα, του ανθρω... Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Όταν αυτή η αλήθεια, αυτές οι πληροφορίες μα φτάνουν, ποιε είναι οι δυνατότητε να βοηθήσουμε εμείς. Ε, στη Σλοβενία, στη χώρα μου, σήμερα το κεντρικό νέο στα στις εφημερίδες είναι το, είσαστε εσείς. Δηλαδή ότι οι ακτιβιστέ του Memorial πήραν το βραβείο Ζαχόρευ. Όλε οι Εφημερίδε το λένε στη χώρα μου, Όμω στην Ρωσία δεν ξέρω πόσε Εφημερίδε θα το αναφέρουν. Και όλα αυτά τα στοιχεία που συζητάμε είναι πολύ ενδιαφέροντα, μα βοηθούν στη δουλειά μα και οι μελέτε που κάνουν από ειδικά όργανα του, που γίνονται από ειδικά όργανα του Κοινοβουλίου είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρέ μελέτε που μα δίνουν ακριβώ ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Επί τη ουσίας, ποια είναι η, δι, η, η, η διάδοση αυτών των πληροφοριών ωστόσο στη Ρωσία και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς έτσι ώστε οι Ρώσοι να παίρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Πριν από 20 χρόνια όταν εμείς στη Ιουκοσλαβία τότε αντισταθήκαμε στον Σταλινισμό Θελήσαμε να μάθουμε, μπορέσαμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες και αυτό συνέβαλε στον να αλλάξει κοινή γνώμη, ο, το, ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει. Και έτσι οι αρχές που είχαν ε, με αυταρχικό τρόπο αρπάξει την εξουσία ε, την έχασαν. Αυτές οι δολοφονίες μου θυμίζουν κάπως τη ρύθμιση λογαριασμών της ε, μαφίας. Δηλαδή, οφθαλμός οφθαλμού και ε, δόντα διοδόντος. Ευχαριστώ. Σύντομα για τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας που γίνεται αναεξάμεινο. Ο διάλογος αυτός, όπως διεξάγεται, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας ημών των Ευρωπαίων. Δεν είναι πραγματικός γνήσιος διάλογος. Και όπως εξήγησαν και οι βραβευθέντες, δεν εξυπηρετεί ούτε τους υπεραφιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χρειάζεται βέβαια ρεαλιστικές αλλά ξεκάθαρες λύσεις και να συμμετάσχουν και οι μη κρατικέ οργανώσει. Όσο ο διάλογο διεξάγεται μεταξύ αξιωματούχων τη Ένωση και αξιωματούχων τη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν θα αποδίδει. Η κυρία Στρίφλερ ήδη έκανε μια πρόταση. Πρέπει να θεσμοποιηθεί ώστε πριν από το διάλογο να διεξάγονται συναντήσεις με μια συγκεκριμένη ατζέντα των Ευρωπαίων αξιωματούχων με τις μη κρατικές οργανώσεις της Ρωσίας. Το ίδιο και μετά τον διάλογο, ώστε να γίνεται αξιολόγηση των διαλόγων. Και τα θέματα που εγγράφονται στην ατζέντα να αφαιρούνται πλέον μόνο εάν οι μη κρατικέ οργανώσει πουν μάλιστα έχει καλώ, δίνουμε πράσινο φω. Έχει δηλαδή λυθεί ένα πρόβλημα όπω θεωρούσαμε και εμεί σωστό. Από τη δική μα σκοπιά πρέπει δε να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο διάλογο αυτό για να επιταχύνουμε τη διαδικασία όπως είπε και ο κ. Στάλερ. Ευχαριστώ κύριε Νόιζερ. Αυτή η συζήτηση ανάμεσα στους υπαλλήλους των ΕΕ και των ΜΚΟ υπάρχουν ε, διάλογοι. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά που εμείς συζητάμε και μεταξύ μας δεν αντικατοπτρίζονται στις διασκέψεις κορυφής. Το θέμα είναι αν μπορούν να γίνουν αυτές οι προματεύσεις ε, και οι διάλογοι στη Ρωσία. Όμως οι ρωσικές αρχές αυτό το έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής ε, καθολικά, ε, μάλλον κάθετα. Ίσως να έχουμε κάποιες περισσότερες ευκαιρίες. Ο Μίνσκι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το βραβείο Ζαχάροφ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ύψη σημασία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω όμω κάτι. Λέτε πω αντιπροσωπεύετε την κοινωνία των πολιτών. Τι είναι η κοινωνία των πολιτών, πόσοι από εσά βρίσκεστε μέσα στην κοινωνία των πολιτών, τι είναι αυτή η κοινωνία των πολιτών, ποιο σα υποστηρίζει. Δεν έχω ακούσει τίποτα ε, ω προ αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, ε εδώ το Κοινοβούλιο είναι εκλεγμένο δημοκρατικά. Έχει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Και γι' αυτό και συνομιλούμε με το Κοινοβούλιο της Ρωσίας. Είπατε όμως πως αυτό δεν είναι νόμιμο το Κοινοβούλιο και ότι όλα αυτά είναι ε, μια εικονική κατάσταση. Εμεί όμω έχουμε επαφέ μαζί του και έχουν αναγνωριστεί οι εκλογέ στη Δούμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λοιπόν την ερώτηση γιατί η κοινωνία των πολιτών δεν είναι πρόθυμη να θεσπίσει τέτοιε δυνάμει στην ε, Ρωσία που να προστατεύουν τα δικαιώματα των ε, ψηφοφόρων και των βουλευτών της Δούμα. Εγώ έρχομαι από την Νότιο Κάφκασο, έχω πάει πολλές φορές εκεί και μάλιστα υπηρέτησα εκεί ως αξιωματικός. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην, στο, στο βόρειο συγγνώμη, Κάφκασο και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πει ότι μπορεί να τα τακτοποιήσει την κατάσταση εκεί εκτός από τη Ρωσία. Εγώ έχω πάει, τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Εσείς μιλάτε για το Βόρειο Κάφκασο. Αλλά τι γίνεται με τον Μπουντόνοφσκ, ε, τον Όστ, αυτούς τους θεωρείτε δολοφόνους. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τη μία πλευρά και με διαφορετικά μέτρα και σταθμά να κρίνουμε την κάθε πλευρά. Πρέπει να ξέρουμε πόσο κόσμο σα στηρίζει. Τι εννοείται όταν λέτε κοινωνία των πολιτών, γιατί στο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας υπάρχουν πολλά κόμματα. 36 κόμματα αντιπροσωπεύονται στο Ρωσικό Κοινοβούλιο. Εάν δεν θεωρείτε πως αυτό είναι ένα γνήσιο κοινοβούλιο, δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε επαφέ τότε μαζί τους. Ε, <clears throat> ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι τις θερμές μου ευχαριστίες για όλα όσα κάνετε, για το σύνολο του έργου σας. Και σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό και σας συγχαίρω θερμά και για το βραβείο Ζαχάροφ. Πρόσφατα αναφέρθηκε αναφέρθηκατε στην σφαγή του Κατίν και υποσχέθηκαν ότι θα γίνει έρευνα χωρίς κανένα περιορισμό. Έγινε αυτό. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί για την ώρα να επανέλθει σε ένα λόγο του Μετβιέντεφ που μίλησε για εξυγχρονισμό της κοινωνίας και δεν ακούν δεν ακούν την μετάφραση Τώρα ακούν. Ωραία. Επανελαμβάνω την ερώτηση. Ο, Πούτιν είχε υποσχεθεί την 1η Σεπτεμβρίου στην Πολωνία έρευνα για την σφαγή του Κατίν χωρίς καμία, κανένα περιορισμό. Και δεύτερο, για την συμφωνία εκτός από το κεφάλαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων για τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας τι άλλο θα περιληφθεί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του Γοντορκόφσκι για την γενεά M. Και αν το διαβάσετε θα μπορέσετε και εσείς να καταλάβετε κύριε Μίσκη τι ακριβώς σημαίνει ε, ε, κοινωνία και μη κρατικέ οργανώσεις στη Ρωσία. Η Γκόμης. Εγώ προέρχομαι από την Πορτογαλία και έχω ζήσει 21 χρόνια υπό δικατορικό καθεστώς. Κατά τη διάρκεια αυτού του καθεστώτος υπήρχε κοινοβούλιο, αχυρένιο με ένα μόνο κόμμα και έπειτα με διάφορα κόμματα. Αλλά ήταν ένα ψευδοκοινοβούλιο που δεν είχε καμία σχέση με την κοινωνία των πολιτών που όπως τώρα μπορεί να εκφραστεί μετά το 1974. Ο κύριος που μίλησε πριν και δεν ξέ, πως δεν ξέρει τι είναι η κοινωνία των πολιτών, να σας πω εγώ ξέρω τι είναι και ξέρω τι θα πει να έχεις κοινωνία των πολιτών που δεν αντιπροσωπεύεται στο κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς θέλω να ρωτήσω τους φίλους και προσκεκλημένους του Is Memorial. Πώς μπορούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουμε την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Εγώ πιστεύω, αν αντλήσω από τη δική μου εμπειρία, ότι το πιο βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών είναι η ενημέρωση, η δωρεάν, η ελεύθερη μάλλον ε, ε, ενημέρωση, η ελευθερία του τύπου. Και ως προς αυτό θέλω να σχολιάσετε ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη πλήση εγκεφάλου που γίνεται από την λογοκρισία και από τα ΜΜΕ, τα ρωσικά, και πώς μπορούμε εμείς στην ε, Ένωση, από δική μας πλευρά δηλαδή, να βοηθήσουμε την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόμες. Τώρα σύντομα ο κύριος Κάσμαρεκ ήθελε να διευκρινίσει κάτι. Αυτά που ανέφερα με τους τετσένους πρόσφυγες στην Πολωνία. Θα ήθελα να ε, διαλευκάνω τα θέματα των Τσετσένων προσφέγων. Έχουν, έγιναν διαδηλώσεις χθες στα πολωνογερμανικά σύνορα σε ό,τι αφορά την παράνομη διέλευση των σύνορων. Από άποψη ανθρωπιστικής κατάστασης δεν πρόκειται να ασκήσει διώξη η Πολωνία για την λαθρεά αυτή διέλευση των σύνορων. Δεν πρόκειται να ασκηθούν κυρώσεις κατά των Τσετσένων. Μάλιστα η Πολωνία είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή σε ό,τι αφορά την, ε, ε, την υποδοχή προσφύγων σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι ότι οι Τσετσένοι δεν θέλουν να παραμείνουν στην Πολωνία. Το χειρότερο πάντως για αυτούς είναι η επαναπρόθεσή τους στην Τσετσενία, γιατί εκεί η ζωή τους απειλείται. Αυτό θα ήταν ε, το χειρότερο σενάριο για αυτούς, ο επαναπατρισμός τους στην Τσετσενία. Σε ό,τι αφορά το Κάτιν, ε, έγινε τον Ιούνιο, τις 7 Ιουνίου συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λίγο μετά τον ε, απολογισμό των θυμάτων από την Πολωνία, τον ακριβή απολογισμό, κατά τη γνώμη της Ρωσίας το έγκλημα αυτό ήταν ένα κοινό έγκλημα. Ε, αυτό, αυτός ο χαρακτηρισμός υιοθετείται από τη Ρωσία και για την ε, δολοφονία της Πολιτκόφσκα. Για απλώς η κλίμακα ήταν διαφορετική. Γιατί τότε είχαμε κοινά εγκλήματα όπου έχασαν τη ζωή τους ε, χιλιάδες άνθρωποι και εδώ έχουμε μεμονωμένα εγκλήματα, κοινά εγκλήματα παρόλα αυτά που χάνουν τη ζωή τους με κάποιοι μεμονωμένοι ακτιβιστές. Πάντω, δυστυχώ από ό,τι φαίνεται, τόσα χρόνια έχουν περάσει και σε ό,τι αφορά τη δολοφονία ανθρώπων, ε, η στάση τη Ρωσία δεν έχει αλλάξει. Έχουμε έξι μόνο λεπτά χρόνο. Θα πρέπει να κάνουμε μια σοφή και δίκαιη κατανομή. Θα πρότεινα δύο λεπτά η κυρία Αλεξέγεβα, δύο λεπτά ο κύριος Ορλόφ και δύο λεπτά στο τέλος ο κύριος Αλμπερτίνη. Κυρία Αλεξέγεβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, υποβλήθηκαν για να τις απαντήσουμε όμως δεν αρκούν δύο λεπτά. Χρειάζεται ολόκληρη διάλεξη. Πολύ ωραία διάλεξη. Και για να σας μιλήσω για την κοινωνία των πολιτών θέλω τουλάχιστον 40 λεπτά. Γιατί κάνω πολύ συχνά διαλέξει με το θέμα αυτό. Είναι δύσκολο λοιπόν να απαντήσω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γνωρίζετε την κατάσταση στον Κάφκασο την ακούτε από τα μάθη και από το πρίσμα ενός Ρώσου αξιωματικού. Γνωρίζουμε αυτή τη θέση και πολλοί την εστερνίζονται. Πολλοί συμπατριώτες μου έχουν την ίδια άποψη. Αντιμετωπίζοντας τα πράγματα υπό το πρίσμα αυτό και στην Τσετσενία υπάρχουν πολύ περισσότεροι στρατιωτικοί και αξιωματικοί του στρατού παρά ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυσικά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο μέσα σε δύο λεπτά. Συγχωρήστε με, αλλά μόνο αυτά μπορώ να σας πω. Μην αισθάνεστε ε, δυσάρεστα, ούτε ενοχή. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ο κύριος Ορλόφ. Σας είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ τον κύριο Μίρσκης για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του. Γιατί δεν υπάρχει πολιτοφυλακή στην Ρωσία, για παράδειγμα, για να ελεχθεί η διεξαγωγή των ελεύθερων και ανώθευτων εκλογών. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι στη Ρωσία, γίνονται εκλογές, αλλά ο νέος εκλογικός νόμος απαγορεύει την παρακολούθηση των εκλογών ε, από μη πολιτικές δυνάμεις. Οπότε ανεξάρτητοι παρατηρητές δεν μπορούν ε, να παρακολουθήσουν τις εκλογές. Φυσικά αν είχα και εγώ ένα δεκάλεπτο και θα μπορούσα κάλλιστα να σας εξηγήσω πώς ανεξάρτητα κόμματα και ανεξάρτητοι παρατηρητές εμποδίζονται στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν τις εκλογές. Σας υπενθυμίζω και τις τελευταίες εκλογές που δεν ήταν κοινοβουλευτικές, δεν ήταν βουλευτικές, ήταν ε, δημοτικές εκλογές. Υπήρξε μία έξαρση δυσαρέσκειας στις τελευταίες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, γιατί ο κόσμος ε, γνωρίζει ότι υπάρχουν καταχρήσεις και νοθείες. Και το θέμα της τρομοκρατίας. Σίγουρα η τρομοκρατία είναι μείζον κίνδυνος για τη Ρωσία και θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Αυτό το επισημαίνουμε και εμείς στην έκθεσή μας. Δεν μπορούμε όμως να καταπολεμήσουμε την κρατική τρομοκρατία που αυτή είναι που σοβεί στη Ρωσία πρώτα απ' όλα. Η κρατική τρομοκρατία που είναι απάνθρωπη και καταπατά όλα τα δικαιώματα είμαστε ανίσχυροι, ανήμποροι απέναντι. Δεν υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσουμε την κρατική τρομοκρατία και αυτή η κρατική τρομοκρατία δρά στη, στη και στο Βόρειο Κάφκασο. Και δυστυχώ είμαστε πολύ ανταπαραγωγικοί στην καταπολέμησή της. Τώρα, αν θα ανοίξουν τα αρχεία και θα εξασφαλιστεί πρόσβαση των ιστορικών σε αυτά, Δυστυχώς όλο και περισσότεροι περιορισμοί ισχύουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα αρχεία. Τώρα πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Αν διαβάσετε τις συστάσεις μας από τη Στοκχόλμη, θα βρείτε συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε να λάβετε για να υποστηρίξετε την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Ορλόφ. Ο κύριος Αλμπερτίνη τώρα. Τι γίνεται, ποιο είναι το συμπέρασμά σα για το κοινό μας έργο στη εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά σε λίγα λεπτά. Όταν πρέπει κάτι να ακούσουμε και να πούμε, δεν χρειάζονται περισσότερα για να επιβεβαιώσουμε το μεγάλο ενδιαφέρον που όλοι μας τρέφουμε για τις προτάσεις και τις ε, συμβουλές που μας δώσατε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε. Μας δώσατε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις, επισκέψεις στους κρατούμενους ε, πολιτικούς αντιρρησίες ε, που είναι απαράδεκτο πράγμα για μια δημοκρατική κατάσταση. Ε, βοήθεια στις οικογένειες ε, για τις ε, θεωρήσεις ώστε να προστατευτούν από τις πιέσεις συστάσεις της Οκχόλμης όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, η βοήθεια στους πρόσφυγες, η οικονομική ανάπτυξη στον Βόρειο Κάφκασο που μπορεί να βοηθήσει στο να αποδυναμεθεί η, αυτή η πρόσφορη κατάσταση για την τρομοκρατία. Ε, υπάρχει μια νέα ε, πολιτική που ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου. Οι, σχέσεις, η, η εταιρική σχέση ανάμεσα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τη σημερινή ε, ε, κοινοπολιτεία, ρωσική κοινοπολιτεία, ε, νομίζω πως ε, είναι παλιά και βασιζόμαστε σε συμφωνίες ε, συνεργασίες που προβλέπει και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν από κάποιες μέρες συμμετείχα σε μια διάσκεψη στην πόλη μου, το Μιλάνο, με τον τίτλο από την κατέρευση του τείχου του Βερολίνου στη συνθήκη της Λισαβόνας. Να λοιπόν σήμερα άκουσα αυτό που μπορεί να συμβεί και ακόμα πρέπει να συμβεί. Ο κομμουνισμός κατέρευσε με το τείχος του πριν από 20 χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει καθιερωθεί η δημοκρατία στους χώρους εκεί όπου άνθεσε αυτή η δικτατορία. Σήμερα όμως υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να, ζήσει ένα, να δώσει μια νέα διάσταση στο ρόλο της και να τοποθετηθεί ως ε, πρωταγωνιστικός συνομιλητής ε, για τα όσα εσείς επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσετε, θα τις χρησιμοποιήσουμε και θα σταθούμε δίπλα σας για τη δημοκρατία στη χώρα σας και από εκεί για την ε, επέκτασή της ολόκληρη τη, τη γη, έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Στρίφλερ. Ναι, κανονικά είχα ακόμα ένα λεπτό. Σα ζητώ μόνο 30 δευτερόλεπτα, γιατί ξέρω πως δεν έχουμε χρόνο. 30 δευτερόλεπτα. Και εγώ θα τα εκμεταλλευτώ για να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία σε σχέση με το διάλογο ανάμεσα στους βουλευτές, τις αρχές, τις επιτροπές και τις ενώσεις. Πραγματικά επιμένω πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να πιστεύετε πως ε,